Ποιότητες, όχι. Εγκρίνονται λοιπόν. Έχουμε την γραπτή δήλωση 29-2010 από τους βουλευτές Τιτσιάνο Μούτη και Άννα Ζαμπόρσκα για την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος γρήγορης ειδοποίησης κατά των παιδοφίλων και της ε, σεξουαλικής παρενόχλησης έχει υπογραφεί αυτή η δήλωση οπότε συγχαίρω τους ε, συναδέλφους οπότε σύμφωνα με το άρθρο 123 του κανονισμού θα δημοσιευτούν στα κείμενα που οποία ε, σε αυτή τη σύνοδο μαζί με τα ονόματα όσων έχουν υπογραφεί